προσεκτικά, καθώς και οι νέες πρωτοβουλίες, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη ενός νέου συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο το πρωί στις 11 Ιουνίου 2013 από τις 8.30 έως τις 2 και από τις 3 ως τις 11 με την ημερήσια διάταξη όπως έχει δημοσιευθεί και την οποία μπορείτε να